Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας και προς μεγάλη χαρά όλων έχει καταφτάσει και η κυρία Ματέρα. Θα περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιδοτικά συστήματα στην Ένωση. Η Επιτροπή Απασχόλησης είναι η καθηλιαρμόδια επιτροπή πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και από πλευρά ισότητα των δύο φίλων ε, Η κυρία Ματέρα είναι η υπεύθυνη, η συγγήτρια η βιωσιμότητα των συνταξιδοτικών συστημάτων αναδείχθηκε σε σημαντικότατο θέμα για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και στην έκθεσή σας εστιάζεται και ε, στην ισότητα των δύο φύλων στα πλαίσια των ε, συνταξιδοτικών συστημάτων. Η διακριτική μεταχείριση που ενδέχεται να υποστούν οι γυναίκες στα πλαίσια του συνταξιδοτικού συστήματος είναι η επίπτωση της μιας πραγματικότητας ότι δηλαδή έχουν εργαστεί για μικρότερο χρονικό διάστημα οι γυναίκες. Επίσης ορισμένα συστήματα λαμβάνεται η υπόψη το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής των γυναικών. και τα συνταξιωτικά συστήματα είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε όταν έχει κάποιος χαμηλότερη αμοιβή πλήττεται φυσικά και λαμβάνει και χαμηλότερη σύνταξη. Προσβλέπουμε στην παρουσίαση της κυρίας Ματέρα που είναι η συγγήτρια όπως λέγαμε για αυτή την έκθεση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη από τους συναδέλφους ε, για την καθυστέρησή μου, αλλά ε, πραγματικά το χιόνι μπλοκάρισε πάρα πολλά αεροδρόμια ε, και υπήρχε κίνδυνος να μην έρθω καθόλου σήμερα. Όπως είπε λοιπόν ήδη η Πρόεδρός μας, αυτό που έχει σχέση με τα πιο κατάλληλα συνταξιωτικά συστήματα, αυτά που θα μπορούν να είναι βιώσιμα. Το όλο θέμα είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβουλίο μας. Και εγώ ε, θεωρώ ότι ανέλαβα μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Με ενδιέφερε πάρα πολύ μάλιστα ε, η ενασχόληση με αυτό το θέμα. Ε, σήμερα λοιπόν ε, ήθελα πάση θυσία να είμαι εδώ, αγωνίστηκα με τα αεροδρόμια και με το χιόνι, γιατί ήθελα να ακούσω την άποψή σας ε, και ήθελα να ακούσω και την άποψη των σχεδόν εισηγητών. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο και παρέστην στην συνάντηση που υπήρξε στην Επιτροπή Απασχόλησης με όλους τους εισηγητές από τις διάφορες επιτροπές και έτσι λοιπόν όλοι μας εστιάσαμε την προσοχή μας στο κατά πόσο είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν τα συνταξιδοτικά συστήματα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η εισηγήτρια η κυρία Όμεν Ρόιτεν απέδωσε μεγάλη σημασία στο θέμα που κυρία Πρόεδρε ε, αναφερθήκατε, αναφέρατε κι εσείς, δηλαδή στις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην εργασία τους και κατόπιν τούτου και στο ότι είναι πολύ δύσκολο να δεχθεί κανείς ε, τι ε, χαμηλότερες συντάξεις, διαφορετικά συνταξιδοτικά συστήματα από αυτά των ανδρών, διότι βεβαίω μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες είναι πολλές φορές αναγκασμένες να δεχτούν μερική απασχόληση ή επισφαλή μορφή εργασίας. Οι γυναίκες υφίστανται συνεχώς διακριτική μεταχείριση. Η συνάδελφος κυρία Όμεν Ρόιτερ μας επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί το σύστημα. Υπάρχει μια μικρή αναφορά στην Πράσινη Βίβλο όπου γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα ύπαρξη σε ισότιμων συνταξιωτικών συστημάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή δικό μας καθήκον είναι να καταθέσουμε τη βέλτιστη δυνατή γνωμοδότηση. Όπως σας είπα, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω αδιακρίτως όλες τις συναδέλφους που έρχονται από τις διάφορες πολιτικές ομάδες γιατί πραγματικά μου κατέθεσαν θαυμάσιες τροπολογίες οι οποίες μου επέτρεψαν να σκεφτώ, να σκεφτώ σε βάθος και θέλω να σας πω ότι από τις 89 τροπολογίες που κατατέθηκαν για αυτή τη γνωμοδότηση, ε, για τις τέσσερις βασικές παραγράφου της γνωμοδότησης, πολλές από αυτές τις τροπολογίες δεν μπορώ δυστυχώς να τις δεχτώ, διότι είναι πέρα από τις αρμοδιότητες και από την ευθύνη που μου ε, εκχωρήσατε. Θα ήθελα ενδεικτικά να αναφέρω μία τροπολογία. Νομίζω ότι η συνάδελφος κυρία Τόμσον δεν είναι παρούσα, διότι... Μισό λεπτό η τροπολογία υπαριθμών 63 της κυρίας Παλιαδέλη όπου καλούνται τα κράτη-μέλη να εισάγουν τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες με ε, συστήματα υποστήριξης ε, στην παιδική ηλικία και άλλα ολοκληρωμένα συστήματα που θα έχουν ως στόχο να περιορίσουν το βάρος ε, που πέφτει στους ώμους των γυναικών οι οποίε καλούνται να μεριμνήσουν και για τους ηλικιωμένους και για τους ασθενείς. Είναι μια πολύ ε, σημαντική έννοια, αλλά ξέρετε, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν μπορεί να ε, συμπεριληφθεί σε αυτή τη γνωμοδότηση, γιατί αν το κάνουμε αυτό υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε τελείως εκτός πεδίου της ε, πρόταση αυτή. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν μου ζήτησε να καταθέσω μια γνωμοδότηση που να είναι πλούσια σε νόημα, σε κίνητρα και όθηση προ τα εμπρός, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε σε άλλα πεδία και να επιμείνουμε, γιατί η διακριτική η μεταχείριση των γυναικών σε αυτό τον τομέα είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στις ε, συναδέλφους, κυρίως ε, σε ορισμένες ε, σκιώδεις ηγήτρες που είναι παρούσες για να μου διευκρινίσουν κάποιες από τις τροπολογίες που εγώ τις χαρακτηρίζω ως εκτός θέματος. Και βεβαίως με χαρά θα ακούσω τη δική τους την άποψη. Ευχαριστούμε. Η κυρία Πλάμπ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου συγχαίροντας πρώτα την εισηγήτρια. Την συγχαίρω για το σχέδιο έκθεσης. Είμαι σκιώδης ε, εισηγήτρια όσον αφορά την ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών SD. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια, αν επιτρέπετε. Φυσικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Έχουμε συζητήσει για αυτό το θέμα και την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και με την Επιτροπή Απασχόλησης τα σχετικά. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής επειδή αναφέρατε πιο πριν το χιόνι, εντάξει. Θα με ικανοποιούσε ιδιαίτερα να βρίσκαμε λύσεις όσες, τόσες λύσεις όσες ε, και ε, τις νυφάδες ε, χιονιού που έπεσαν τις τελευταίες μέρες. Πολλές λύσεις λοιπόν. Αν θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να ε, συγκροτήσουν κάποια μέτρα για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Επανέρχομαι στην έκθεση και αυτό που προσπάθησα είναι να γίνει λόγος, να κάνουμε λόγο για την προαγωγή της ελαστικότητας κάποια ελαστικότητα όσον αφορά τον καθορισμό των ηλικιακών ορίων, λαμβάνοντα πάντα υπόψη τη διάσταση του φύλου. Δεν νομίζω ότι η αύξηση όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά όρια θα είναι η καθοριστική τελεσίδικη λύση για τα δημογραφικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Υπάρχουν όμως κάποιες μελέτες που αποδεικνύουν ότι η αύξηση, μια αύξηση στην ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών θα μπορούσε πιθανώς να οδηγήσει σε μια αύξηση, αύξηση του αριθμού γυναικών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων γυναικών που θα γίνονται όλο και πιο φτωχότερες και θα απειλούνται από τη φτώχεια. Η φτώχεια λοιπόν μεταξύ των γυναικών θα μπορούσε να αυξηθεί αν ακολουθηθεί αυτή η λογική. Ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να παγιώσουν ένα επαρκή χαρακτήρα συντάξεων, καταπολεμώντας την αρνητική διάκριση εις βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα μειώνοντας το μισθολογικό χάσμα, τη μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα ελάχιστο 10% που το 2020 θα πρέπει να έχει μειωθεί όσον αφορά τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών γυναικών. Επίσης έγινε λόγος για τις περιόδους που ανάλωσαν γυναίκες και άνδρες μεριμνώντας και περιθάλποντας παιδιά ή ηλικιωμένους στο σπίτι, στην οικογένεια. Θα έπρεπε να αναγνωρίζεται αυτή η περίοδος, αυτή η χρονική περίοδος ε, με τη μέθοδο υπολογισμού ως ενεργός περίοδος ε, για να μπορούν να αναγνωριστούν για την συνταξιοδότηση και για την, ας το πω έτσι, αντιστάθμιση αυτής της ε, εργασίας. Ακόμα και αν η κυρία Λούλινγκ με μια τροπολογία με ρημνά για δύο χρόνια περίοδο που θα καλύπτεται, που είναι η περίοδος που οι άνδρες και οι γυναίκες προσέχουν τα νεογνά και τα βρέφη, με ρημνούν για αυτά, θα ήθελα να ξεκινήσει μια διαδικασία για τη διαγραφή, την κατάργηση του άρθρου 5 στην παράγραφο 2 της οδηγίας 113 του 2004 όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που επιτρέπει αρνητική διακριτική μεταχείριση εις βάρος των γυναικών όσον αφορά και τις συντάξεις της ίδιας. Ταυτόχρονα ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει μια μελέτη όσον αφορά τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων των συνταξιοδοτικών συστημάτων στην ίδια τη ζωή των γυναικών και τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή των γυναικών λαμβάνοντας υπόψη τους εξής στόχους. Την εξατομίκευση των δικαιωμάτων συνταξιοδότηση και συντάξεως καθορισμό μηχανισμών που θα καθιστούν εφικτή την αντιστήχηση των αναγκών με τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας. Ιδιαίτερα όταν γίνεται λόγος για την μέρημνα και την φροντίδα εξαρτώμενων, εξαρτημένων ατόμων στην οικογένεια παιδιών, υπερήλικων και ιδιαίτερα όσον αφορά την ένταξη στον τρίτο πυλώνα με τις διάφορες ανάγκες για τις διάφορες ομάδες γυναικών όπως μετανάστριες γυναίκες ή εκείνες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες ή τις γυναίκες με ειδικές ανάγκες, με αναπηρίες. Ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι αναγκαίο τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν την έρευνα των επιπτώσεων διαφορετικών τύπων που χρησιμοποιούνται σήμερα για τον υπολογισμό και τους δείκτες όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας σε προχωρημένη ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παραμέτρους. Καλό επίσης καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, κάνει μια σφαιρική συνολική αποτίμηση των επιπτώσεων στις γυναίκες όλων των νέων μορφών και τύπων που έχουν εισαχθεί με τις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Καλούνται επίσης τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τους όρους και προποθέσει εργασία και να δώσουν κίνητρα επίση για τι γυναίκε, να παραμένουν οι γυναίκες επί επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο, στην εργασία τους εφόσον το επιθυμούν λαμβάνοντας πάντα υπόψη την πτυχή του φίλου. Ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι η αύξηση του ορίου ηλικίας για την συνταξιοδότηση θα έπρεπε να είναι εθελοντικού, εθελούσιου χαρακτήρα και όχι δεσμευτική, όχι υποχρεωτική. Επίσης καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τις πιέσεις επί των κρατών μελών για την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων κρατικών συστημάτων συνταξιοδότησης συνταξιοδοτικών συστημάτων. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει ένα κρατικό σύστημα δημόσιου χαρακτήρα που θα διέπει τις συντάξεις. Εγώ θεωρώ ότι ο πυλώνας 1, ο πρώτος πυλώνας είναι ο καλύτερος για αυτή τη δουλειά, διότι διασφαλίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και άρει τις ε, διαφορές και τις αρνητικές διακρίσεις. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις ε, που θα είχα να κάνω και που μπορούν, μπορεί να βρεθούν στις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για αυτό το θέμα. Και φυσικά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα συζητήσουμε φυσικά με την κυρία Ματέρα που θα έρθουμε σε επαφή μαζί της για την θέση αυτή που έχουμε. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Κορνέλη, τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή μου θυμίζει ε, το 1996 όταν προτέπησα δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ε, σύμβουλος για πολιτικά θέματα. Και τότε στην Επιτροπή ε, Δικαιωμάτων Γυναικών είχαμε μια πρόταση για το συνταξιδοτικό και τότε ε, θελήσαμε να λάβουμε υπόψη στο γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Ε, κρίναμε ότι αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να εξαλειφθεί. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε επί του θέματος με έντονο ύφος, αλλά δυστυχώς το Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση του Κοινοβουλίου και δεν έγινε τίποτα. Βεβαίως δεν ήταν εύκολο να συζητήσει κανείς αυτά τα θέματα, διότι είτε τίποτα δεν γινόταν τότε στα συνταξιωτικά συστήματα και γενικότερα στις ε, συντάξεις ε, είτε για άλλους ε, λόγους βούλησης. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν στο συνταξιοδοτικό. Διανύουμε περίοδο ή θα αντιμετωπίσουμε κρίση μετά από 10 χρόνια που η κρίση αυτή θα είναι πολύ χειρότερη από την τρέχουσα. Γι' αυτό λοιπόν αν ε, θελήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα ίσως ε, θα πρέπει να εξαλείψουμε και τα τελευταία στοιχεία ε, διακριτικής μεταχείρισης που υπάρχουν. Τροπολογία υπαριθμών 32 της κυρίας Τόψον. Εγώ τη στηρίζω ανεπιφύλακτα. Είναι καλύτερη ακόμα και από τη δική μου επί του ιδίου θέματος. και έτσι λοιπόν αντιμετωπίζονται θέματα που ήδη θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε να εξετάσουμε το 1996. Να μην υπάρχει διάκριση βάρο των γυναικών επειδή έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωή. Επίση, να διασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να καταργηθούν τα πλεονεκτήματα ε, των ανδρών ε, που έχουν ειδικά ε, δικαιώματα και κανείς δεν θα πρέπει να αποκλείεται από σύνταξη είτε δουλεύει με μερική απασχόληση είτε με άτυπη μορφή εργασίας είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Θα ήθελα λοιπόν να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία και στη θέση των μεταναστριών. Η τροπολογία υπερθμών 47 ακριβώς αυτό το θέμα εξετάζει. Πρέπει βέβαια να είμαστε προσεκτικοί να μην αφαιρέσουμε τα κίνητρα των γυναικών για να εργαστούν. Ε, η δουλειά να κατανέμεται ισότιμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και να μην προσφέρουμε στις γυναίκες όλους εκείνους τους λόγους που θα τις αναγκάσουν να παρατηθούν από οποιαδήποτε μορφή εργασίας. Πρέπει τα επόμενα χρόνια να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Ένα τελευταίο θέμα. Η κυρία Πλάμ αναφέρθηκε στον πρώτο σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα. Γνωρίζω ότι εδώ πρόκειται για μια τεράστια συζήτηση. Εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συμφωνήσουμε επ' αυτού, γιατί ε, πρόκειται ε, για κάτι που εμπίπτει αναμφίβολα στις εθνικές αρμοδιότητες. Στην Ολλανδία έχουμε ένα ισχυρό ε, συνταξιωτικό δεύτερο πυλώνα. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα ε, των συντάξεων, αλλά είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι οι συντάξεις του δεύτερου πυλώνα ε, θα διατίθενται σε όλους και δεν θα υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Σας ευχαριστούμε, κυρία Λούλιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω συντάξει και εγώ κάποιες ε, τροπολογίες που έχουν ε, ως στόχο να ε, διασαφηνίσουν την κατάσταση και να είμαστε και πιο συνεκτικοί. Πρώτον, τροπολογία για το εκτιμώντας την αιτιολογική σκέψη 1, διότι άλλο υπολογισμός των συντάξεων Και άλλο αναλογιστικό ε, υπολογισμός ε, πρέπει να μεριμνήσουμε το ώστε να υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση των συνταξιδοτικών συστημάτων και υπέβαλα αυτή την τροπολογία. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε ε, τα σίκα με τα μήλα. Επίσης, για το ε, εκτιμώντας β, έχω υποβάλει μια τροπολογία γιατί είναι σημαντικό να ε, υποδείξουμε ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες σε σχέση με τους άντρες να πάψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή να ε, ε, μην εργάζονται, να μην έχουν συμβάσει σε πλήρους ωραρίου όπως οι άντρες ε, και αυτό επηρεάζει τη σύνταξή τους ε, στην ε, χώρα μου. Έχουμε μία αντιστάθμιση, την ονομάζουμε baby years, τα χρόνια των νεογνών. Δηλαδή, ανά παιδί υπολογίζονται δύο χρόνια για τα οποία αντισταθμίζεται η απώλεια της σύνταξης των γυναικών και νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μα σε τέτοιου είδου αιτήματα που είναι λογικά, μέτρα που ήδη υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη και να μην ζητάμε να χορηγηθούν συντάξει σε κάποιου που ποτέ δεν εργάστηκαν ε, ή που δεν είχαν ε, συμβάσει πλήρου χρόνου euh, euh, ε, που είχαν μερική απασχόληση ε, ε, γιατί ε, τα περισσότερα συστήματα βασίζονται στις εισφορές αλλά άλλα βασίζονται στο μισθό. Δεν μπορείτε να δώσετε σε κάποιον άντρα ή γυναίκα μία αυξημένη σύνταξη γιατί είχε χαμηλότερο μισθό ή γιατί δεν εργάστηκε όλο το χρονικό διάστημα οι άντρε έχουν ε, πιο πλήρε επαγγελματικέ ε, σταδιοδρομίε. Όσοι έχουν εργαστεί για 40 χρόνια και έχουν καταβάλει τι εισφορέ ε, στου εργοδότε του, εντάξει, και σε εμά το κράτο καταβάλει τη σύνταξη. Είναι λογικό λοιπόν να έχουν αυτή αυξημένη σύνταξη σε σχέση με αυτού που είχαν σύμβαση μερική απασχόληση. Δεν μπορείτε να το αντισταθμίσετε αυτό με οποιοδήποτε σύστημα συνταξιωτικού συστήματο γιατί θα ήταν άνισο ενώπιον αυτών που έχουν καταβάλει ψηλό περισσότερες εισφορές. Οπότε ε, θα πρέπει να διαρευνήσουμε αυτή την ιδέα, δηλαδή αντιστάθμισμα σε σχέση με αυτά που σας είπα, τα baby years, ε, ε, τα χρόνια που σταματάει η γυναίκα τη δουλειά για να φροντίσει τα παιδιά ή για να φροντίσει κάποιον άλλον που το χρειάζεται στην οικογένεια. Υπάρχουν άλλα πράγματα βέβαια που δεν είναι συμβατά με τα ε, συστήματα και σας λέω ότι κάποιες ρυθμίσεις θα ήταν άνισες και θα βάριναν άλλους ασφαλισμένους ε, ε, θα ήθελα να διαγράψουμε την, την αιτιολογική σκέψη εσύ, γιατί μιλάμε για τη φτώχεια που πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και τους συνταξιούχους. Μα στη χώρα μου είναι το αντίθετο. Η καλύτερη του χωριού είναι οι συνταξιούχοι. Ε, γιατί έχουμε αρκετά καλές συντάξεις ε, και ε, οι πλέον ευνοημένες είναι οι γυναίκες που ποτέ δεν εργάστηκαν, που παντρεύτηκαν κάποιον που δούλευε όλη τη ζωή του και ακόμα καλύτερα αν δούλευε καθ' όλη τη διάρκεια της ενεργούς ηλικίας του και οι, οι, αυτοί που βρίσκονται στη χειρότερη θέση είναι οι διαζευμένοι και αυτοί που δεν εργάστηκαν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, άνθρωποι της γενιάς μου ας πούμε. Στη χώρα μου καμία γυναίκα που δούλεψε 40 χρόνια όπως εγώ παραδείγματος χάρη και έχει καταβάλει εισφορές ε, για 40 χρόνια ε, ε, δεν έχει τόσο όσο κάποιες χείρες. Ε, ε, ξέρετε, στη δικιά μου την εποχή οι γυναίκες δεν ήταν διευθύντριες, αλλά η χείρα ενός διευθυντή παίρνει τουλάχιστον χίλια ευρώ περισσότερα στη σύνταξή σε σχέση με μένα που έχω δουλέψει <laughs> για 40 χρόνια αλλά αυτό είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε. Δεν πρέπει να αναφέρουμε αυτό το στοιχείο για τις γυναίκες. Το σημαντικό είναι να δούμε πώς θα αντισταθμίσουμε τις περιόδους κατά τις οποίες αφοσιώθηκαν στην ανατροφή των παιδιών τους, στη φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας που το χρειάζονταν και επιμένω, το τονίζω, γιατί δεν πρέπει να υποβάλουμε τέτοια αιτήματα, όπως πολύ σωστά είπε και η συγγήτριά μας, που εκπίπτουν του πεδίου. Ε, ε, μπορεί να ξεκινάνε κάποιες τροπολογίες από καλέ προθέσεις αλλά πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Αν θέλετε να ληφθεί υπόψη το σχέδιο γνωμοδότησης μετά την εγκρίσή του συγκεντρωθείτε στα βασικά ε, στοιχεία, τα, ε, τα σημεία που έχουν σημασία για τις γυναίκες. Άλλο παράδειγμα... Μία παράγραφος που επίσης διαγράφω λέει εκτιμά ότι τα συνδοξιδοτικά συστήματα πρέπει να βασίζονται σε ενδεδειγμένα και βιώσιμα κριτήρια και να λαμβάνουν υπόψη τις, ε, περιο, ε, να λαμβάνουν υπόψη περιόδους μερικής απασχόλησης ε, ή μη εργασίας. Ε, Δεν μπορούμε αυτό, ε, αυτό να μα οδηγήσει σε πλεονέκτημα για τι γυναίκε ή και για του άντρε, γιατί μπορεί οι άντρε να έχουν αναθρέψει τα παιδιά και να έχουν διακόψει ε, τι επαγγελματικέ του δραστηριότητε τα πρώτα χρόνια ζωή του παιδιού του. Οπότε και αυτοί θα έπρεπε να υποφεληθούν όπω και οι γυναίκε. Ε, θα ήθελα λοιπόν να διαγράψουμε όλα αυτά που ξεκινούν σίγουρα από καλέ προθέσει, αλλά πραγματικά καμία σχέση δεν έχουν με το θέμα μα ε, και να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας ε, σε ρεαλιστικές προτάσεις που ενδέχεται να ληφθούν υπόψη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Ματέρα, θέλετε να κάνετε κάποιες καταληκτικές ε, παρατηρήσεις μετά τη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, σημείωσα όλες ε, αυτές τις ε, παρατηρήσεις των συναδέλφων και νομίζω ότι για ορισμένα θέματα συμφωνούμε απόλυτα. Είναι σημαντικό να μην αυξηθεί περαιτέρω η ηλικία συνταξιοδότησης γιατί οι γυναίκες συνεισφέρουν σημαντικά στην κοινωνία Παράλληλα βέβαια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες ε, εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, σε κινδύνους ε, που μπορούν να επηρεάσουν κάλλιστα την υγεία της, τη φυσική της κατάσταση. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ε, μιλάμε στην Επιτροπή για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής ε, των γυναικών, κάτι το οποίο ε, συνεπάγεται και τον κίνδυνο της ε, φτώχειας και της μοναξιάς. Πολλές φορές το έχω επισημάνει αυτό κατά το παρελθόν, ότι δεν πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω η ηλικία συνταξιοδότηση γιατί πολλά κρατημέλη και η ίδια η Ιταλία δεν λαμβάνουν υπόψη τους ε, ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ομοιομορφία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με αυτά που μόλις τώρα είπε η κυρία Λούλινγκ, αναμφίβολα δεν πρέπει να νοθευτεί μία γνωμοδότηση η οποία θα πρέπει να είναι περιορισμένη για καθαρά τεχνικούς λόγους. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε σύγχυση σε όποιον θα διαβάσει την γνωμοδότηση. Πολύ ωραία αυτά που λέγονται ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις μετανάστριες, στις εθνοτικές ομάδες, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην κάνουμε το λάθος να επαναφέρουμε εκθέσεις που υπήρξαν κατά το παρελθόν γιατί στη τελική ανάλυση ε, πρέπει να συμφωνήσουμε σε πράγματα που είναι σημαντικά. Ε, ας συνεχίσουμε λοιπόν να μιλάμε για την ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες δηλαδή για το ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί ε, η διαφορά που υπάρχει στο μισθολογικό. Δεν πρέπει όμως να αναφέρουμε εκεί τα πάντα και, τα, ε, και τους λόγους που υπάρχουν πάρα πολλούς και διαφορετικούς γιατί τελικά κινδυνεύουμε να μην μας λάβουν σοβαρά υπόψη. Σε σχέση με αυτά ε, που είπε η κυρία Κορνέλισεν συμφωνώ και εγώ ότι εδώ πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα ε, το θέμα αυτό υπήρξε και πριν από 10 και ακόμα περισσότερα χρόνια. Αναμφίβολα σήμερα το Κοινοβούλιο χάρη της ε, συνθήκης Λισαβόνας ε, έχει νέες αρμοδιότητες έχει περισσότερη εξουσία. Ας το εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτό για να ακουστεί η φωνή μας. Και η γνωμοδότηση έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, να εισακουστεί η φωνή μας. Κατόπιν, διάβαζα λιγάκι τις σημειώσεις μου. Είναι πολύ σημαντική η τροπολογία της κυρίας Τόμσον που είναι μια νέα τροπολογία όπου ε, λαμβάνει υπόψη της ε, το ότι είναι σημαντικό να μην περιοριστούμε στις συμβάσεις να λάβουμε υπόψη μας σε σχέση με τη σταξιοδότηση όλες τις μορφές συμβάσεων που υπάρχουν. Σωστό είναι αυτό και δίκαιο, αλλά είναι μια ε, διαφορετική, μια τελείως νέα ε, τροπολογία και ίσως ε, τις επόμενες ημέρες αν τελικά και το χιόνι μας αναγκάσει να μείνουμε εδώ θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τροπολογίες θεωρώ ότι ε, πολλές πρέπει να συμπεριληφθούν. Δεν θέλω βέβαια να ξεχάσω τίποτα, αλλά νομίζω ότι προς το παρόν αυτά είχα να πω και αν θέλω να πω αργότερα και κάτι άλλο θα ξαναζητήσω βέβαια το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Στις 13 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Απασχόλησης 1 Φεβρουαρίου, τότε θα γίνει η ψηφοφαρία ε, και το Φεβρουάριο ευελπιστούμε να περάσει η γνωμοδότηση και η έκθεση γνώμη και την Ολομέλεια. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο για σήμερα. Θα αρχίσουμε τώρα τη συνεδρίαση των συντονιστών ε, με κάποια καθυστέρηση. Ελπίζω ταχύτατα να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ πάντως για την συνεδρίαση της Επιτροπής.